Mr. Brons. You're very welcome. okay. Um, I don't want to, uh, to... Δεν θέλω να τιμωρηθούν αυτοί που είναι παρόντες και είναι και στην ώρα τους. Yes. I thought that it would punctuate the silence while waiting for our colleagues to attend. Um, Νομίζω ότι επειδή ο χρόνος μας πιέζει και επειδή άλλοι θα θέλουν να μιλήσουν, θα ήθελα να σας πω το εξής. Αντί να κάνουμε μια ενιαία συνεδρίαση, να μοιράσουμε στις 17, στις, εδώ, στις 18 εκεί και να δούμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν εκφράσει την επιθυμία να πάρουν το λόγο. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο εάν μοιράσουμε και κατανείμουν κατά αυτόν τον τρόπο την συνεδρίαση. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, κάθε φορά που το κάναμε αυτό, ε, ακούω την πρότασή σας, μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα, όμως ο λόγος που το κάναμε είναι ότι έχουμε πολλά θέματα και λίγο χρόνο, γι' αυτό προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τις δύο συνεδριάσεις σε μία. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. επειδή δεν είναι όλοι παρόντες, θα κοιτάξω πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα σημεία για τα οποία οι συγκητές είναι παρόντες, έτσι ώστε να μην περιμένουμε μισή ώρα κάθε φορά και να την συμπτύξουμε κατά κάποιο τρόπο. Καταρχήν, συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη ως έχει. Δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Θα πρέπει να ξεκινήσω με κάποιες συστάσεις όσον αφορά διορισμούς εισηγητών. Χιμένες Μπεσερίλ για την πρόταση οδηγίας όσον αφορά την απόφαση πλαίσιο για την παράνομη εμπορία ναρκωτικών. Η κυρία Αντζελίλη επίσης για την γνωμοδότηση ΦΕΜ πρόκειται για έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τη βία κατά των γυναικών. Επίσης τρίτη συγκήτρια κυρία Ρόιτοβα Πρόκειται τις απαλλαγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η κυρία Ματιού όσον αφορά την απαλλαγή για την προστασία δεδομένων, της υπηρεσίας προστασία δεδομένων Eurojust, European ε, Asylum Support Office, Frontex, Europol για το 2012. Υπάρχουν αντιρρήσεις για τον διορισμό αυτών των εισηγητών. Όχι, θεωρούμε λοιπόν ότι εγκρίνονται. Θα έπρεπε επίσης να σας πω ότι σήμερα δεν υπάρχει διερμηνία στα δανέζικα, φιλανδέζικα, ιστονικά, μαλτέζικα και κροατικά λόγω της, του αριθμού των καμπινών σε αυτήν την αίθουσα. Και μπορούμε να συνεχίσουμε με το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. συγκητής είναι ο κύριος ε, Μωράες. Πρόκειπε για το θέμα της ε, Διαθεσμικής Συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ, Σοφή. Βεβαίως και έχουμε την ε, πρόταση αυτή. Δεν είχαμε χρόνο για να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Έχουμε ένα ε, κείμενο για τους εποχιακούς εργαζόμενους, μετανάστες και βεβαίως εδώ καλύπτονται μετανάστες από διάφορες περιοχές. Περιμένω από τους σκιώδεις εισηγητές. Δεν υπάρχουν πολλά μέλη παρόντες. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν την απουσία τους ως ευκαιρία για να ευχαριστήσω το προσωπικό της Επιτροπής, της Γραμματείας σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την υποστήριξή σας. Πρόκειται για ένα θέμα βεβαίως που προκαλεί έντονες συζητήσεις. Στις 14 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η συζήτηση στην Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η συνεργασία για ένα τόσο λεπτό θέμα ήταν εξαιρετική με τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες και πραγματικά φτάσαμε σε ένα αρκετά πλήρες ε, και αρμονικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους και επαναλαμβάνω θα ψηφίσουμε, συγγνώμη, θα ψηφίσουμε στις 14 Νοεμβρίου. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μπορώ τώρα να σας παρουσιάσω Τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο στις 17 Οκτωβρίου έλαβε χώρα αυτή η τριμερή συνάντηση και πρέπει να σας πω ότι συμφωνήσαμε όσον αφορά τις ε, δύο προτάσεις ε, για κατοξιοδότηση πράξης. Πρόκειται για τα δύο προγράμματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και τα κονδύλια home για τα ειδικά προγράμματα, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα εθνικά προγράμματα. Είναι τελείως ακατανόητο, αλλά σας το διαβάζω όσο έχει. Πρώτη φορά σε ακούω να το παραδέχεστε όμως. Λοιπόν, ο πρόεδρος, ο κύριος Λόπες δηλαδή και όχι εγώ, σας έχει διανύμει την πρόταση που μας έχει ανεπίσημα σταλεί από την Επιτροπή και που βεβαίως στηρίζεται από την Προεδρία, από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλει τις προτάσεις του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μας θεωρεί ότι βεβαίως εδώ θα πρέπει να εξεταστούν όλες τις περιπτώσεις αποκλήσεων, οι οποίες μπορεί να γίνουν δεκτές μόνο εάν δεν ξεπνούν κάποια συγκεκριμένα ποσοστά. Και ο Πρόεδρος μου ζητά να παρουσιάσω τις προτάσεις σας, τα σχόλιά σας, εάν υπάρχουν. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως εξαιρετικά ε, λεπτό. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4. Ο συνάδελφος, ο κύριος Ήλτσεφ, είναι παρόν. Ήδη από τις 18, συγγνώμη, γνωρίζουμε ήδη από το Σεπτέμβριο ότι από τις 18-20 Σεπτεμβρίου, όταν η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έστειλε μια αντιπροσωπεία στη Βουλγαρία και στα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας-Ελλάδας για την εξέταση των θεμάτων αυτών που αφορούν ε, την ε, εμπορία τσιγάρων στα σύνορα αυτά. Ξέρετε ότι υπήρχαν και μέλη της δικής μας Επιτροπής ο κύριος Ήλτσεφ, ο οποίος συμμετείχε σε αυτήν την αντιπροσωπεία, εξ ονόματος λοιπόν της δικής μας Επιτροπής, παρουσίασε μία έκθεση. Ο κύριος Μούλτερ δεν είναι παρόν. Ίσως έχουμε και κάποιο μέλος από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ήλτσεφ. και ο πρόεδρος, ο κύριος Αγγιράρ, αλλά και εγώ σαν αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ήμουν παρόν σε αυτήν την αποστολή. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψή μας εκεί. Ήταν βεβαίως διοργανωμένη από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Και από την αρχή της αύξησης αυτού του κύματος μεταναστών, το πέρασμα από την Τουρκία στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργούν τα διάφορα συστήματα ελέγχου της μετανάστευσης. Και διαπιστώσαμε βεβαίως ότι ο εξοπλισμός, η επενδύσεις, η κατάρτιση του προσωπικού επιτόπου ήταν εξαιρετικά θετική, τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες, διότι αυτό που πραγματικά διαπιστώσαμε είναι ότι ήδη από το τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά και τώρα αυτό έχει αυξηθεί, είναι ένα πολύ σημαντικό και αυξανόμενο κύμα μεταναστών, άτομα τα οποία προσπαθούν να περάσουν από τα σύνορα, από την Τουρκία προς την Βουλγαρία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτά τα κύματα μεταναστών, αντιμετωπίζουν και πάρα πολύ ε, τεράστιες δυσκολίες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, αν θέλετε, μεταναστών. Αυτοί που λένε ότι η προέλευσή τους είναι η Συρία και ξέρετε ότι ο εντοπισμός αυτών των ανθρώπων της προέλευσής τους, καθότι τις περισσότερες φορές δεν έχουν ε, χαρτιά, είναι εξαιρετικά δύσκολη και οι διαδικασίες αργές. Σήμερα ξέρουμε ότι οι διαδικασίες αυτές θα επισπευθούν και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τρεις με τέσσερις ημέρες. Η άλλη κατηγορία είναι πρόσφυγες, μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν απολύτως κανένα έγγραφο έντυπο μαζί τους, δίνουν λανθασμένες πληροφορίες και βεβαίως πολλές φορές διαπιστώνεται ότι κάποιοι από αυτούς έχουν και ε, ποινικό μητρό, εγκληματικές δραστηριότητες Οι περισσότεροι προέρχονται από την Βόρεια Αφρική. Υπάρχουν και κάποιοι που προέρχονται από το Ιράκ, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν. Η Βουλγαρία είναι μια χώρα που δεν έχει εμπειρία αντιμετώπισης τέτοιων κυμάτων μεταναστών και βεβαίως προσπαθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσει παρέχοντας ιατρική περίθαλψη, ανθρωπιστική βοήθεια, στέγη. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το 75% αυτών που επικαλούνται ως χώρα προέλευσης στην Συρία είναι γυναίκες και παιδιά. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των παιδιών είναι και συνόδευτα Και καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές το πέρασμα από την Τουρκία και ξέρετε ότι πρόκειται για διαδρομές που ξεπερνούν τα 1500 χιλιόμετρα ή 2000 χιλιόμετρα από ε, την περιοχή που υπάρχουν τα διάφορα στρατόπεδα, οι καταβλισμοί αυτών των ανθρώπων στο Χατάι μέχρι το βουλγαρικό σύνορο. Διασχίζουν λοιπόν όλη την Τουρκία με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δεν μιλούν οι περισσότεροι από αυτούς τουρκικά, μιλούν ούτε καν αραβικά δεν μιλούν οι περισσότεροι από αυτούς, μιλούν ουρντού ή άλλες διαλέκτους, άλλες γλώσσες. εξωτικές γλώσσες και διαλέκτους μιλών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι αρχές της Βουλγαρίας κάνουν ό,τι μπορούν όπως σας είπα. Έχει προετοιμαστεί μάλιστα και ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα υλοποιηθεί τους επόμενους έξι μήνες με πολύ συγκεκριμένους στόχους αντιμετωπίζουμε προκλήσεις όπως καταλαβαίνετε με τη φύλαξη των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι από αυτούς τους στόχους όπως έχουν προετοιμαστεί σε αυτό το σχέδιο, καταλαβαίνετε είναι ίσως και λίγο αμφιλεγόμενοι. Ο βασικός στόχος είναι να περιοριστεί ο αριθμός αυτών που διασχίζουν τα σύνορα. Και όταν μιλώ για αμφιλεγόμενους στόχους θα σας πω ότι προετοιμάζεται ένας ένας τείχος, ένα τρόπος να περιορίζονται οι διαδρομές και τα σημεία ελέγχου και τα περάσματα από την Τουρκία. Και καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι οποίοι στέλνονται πίσω στις χώρες τους, όχι βέβαια στη Συρία, προς την Τινησία, Αλγερία, Αίγυπτο, Λιβύη, Ιράκ, Ιράν, αυτό βέβαια δεν είναι πάντοτε δυνατόν, με αεροπορικές πτήσεις. Και βεβαίως, όπως σας είπα, υπάρχουν τρομερά προβλήματα επικοινωνίας, ε, αυτοί οι άνθρωποι δεν ομιλούν ε, καμία γλώσσα της περιοχής. Υπάρχει πρόβλημα κατάρτισης ε, και των αρχών που κάνουν αυτούς τους ελέγχους και πρέπει να διαχειριστούν αυτά τα κύματα μεταναστών. Αυτό δηλαδή έχει οδηγήσει στην περιοχή σε πολύ μεγάλες εντάσεις και εθνικές εξάρσεις. Επίσης, όσον αφορά τις συμφωνίες επανεισδοχής ή άλλες συμφωνίες για την διαχείριση, υπάρχει συμφωνία από το 1967 μεταξύ Άγκυρας και Σόφιας, κάτι που βεβαίως σήμερα δεν μπορεί να καλύψει τα σημερινά προβλήματα. Και από την άλλη έχουμε και την ε, έλλειψη προθυμίας ε, της Τουρκίας να υπογράψει την Συμφωνία Επανεισδοχής. Αυτό καταλαβαίνετε αυξάνει τα προβλήματα και η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει ενός είδους διαπραγμάτευση. Ενδεχομένως δηλαδή θα μπορούσε να υπογράψει αυτήν την συμφωνία επανεισδοχής, να στηρίξει, δηλαδή να βοηθήσει τις αρχές ε, της Βουλγαρίας έναντι κάποιας ε, πιο φιλελεύθερης πολιτικής ε, για τις θεωρήσεις ή κάποιο άλλο θέμα το οποίο διαπραγματεύονται. Επίσης πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν δυνάμεις χωροφυλακής στην περιοχή, πεζοί, οι οποίοι προσπαθούν να ρυθμίσουν περιπτώσεις μεταναστών οι οποίοι ουσιαστικά φαίνεται, το γνωρίζουμε διότι είναι εμφανές, ότι καθοδηγούνται από τους ε, τουρκικές ε, δυνάμεις για το πώς να περάσουν καλύτερα τα σύνορα, πώς δηλαδή να μπουν με μεγαλύτερη ευκολία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι έχουν τα πράγματα και ξέρουμε σήμερα ότι αν όλοι αυτοί μπορούσαν να παραμείνουν στην ε, Τουρκία σε ασφαλές ε, ε, περιβάλλον, σε ένα ασφαλή καταβλισμό, προστατευμένοι από τις ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα στη Συρία, ε, δεν θα είχαν ποτέ περάσει, διασχίσει όλη την Τουρκία για να φτάσουν μέχρι τα βουλγαρικά σύνορα. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα δύσκολο θέμα και πρέπει να σας πω ότι και η διπλωματική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας οι επαφές που έχουν με τους Τούρκους ομολογούς τους, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, και η συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων που τώρα σας παρουσιάζω ε, συνεχίζεται. Και βεβαίως ε, η Επίτροπος της Βουλγαρίας ε, συμμετέχει ενεργά και διευκολύνει αυτές τις επαφές. Συζητώντας ε, τις διαφορετικές κατηγορίες ε, μεταναστών, το καθεστώς τους, η προσπάθεια να εξευρεθεί ένας ακριβής ορισμός για το τι είναι μετανάστης, τι είναι οικονομικός μετανάστης, τι είναι πρόσφυγας, τι είναι πολιτικός πρόσφυγας. Όλα αυτά είναι, αν θέλετε, ε, πολύ θεωρητικά, πολύ ρομαντικά. Και στην πράξη πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς πήγαμε επί τόπου και είδαμε την κατάσταση και το θέμα του ασύλου παραδείγματος χάρη είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Αυτό που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι η ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι κάτι που θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Με ενημερώνουν από τη γραμματεία ότι έχει τεθεί στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών αύριο η πιθανότητα να συζητήσουμε μια ε, συμπληρωματική επίσκεψη επιτόπου. Κύριος Μπλόντς. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό για τον έλεγχο των συνόρων. Όμως αυτό φαίνεται ότι δεν αποτρέπει τις μεταναστευτικές ροές, απλώς καταγράφει τους μετανάστες που εισέρχονται. Πριν 18 μήνες είχε έρθει εδώ ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex και μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά σύνορα μας είπε ότι δεν τα ε, διέρχεται κανείς χωρίς να εντοπιστεί. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κρατούνται για λίγο μικρό χρονικό διάστημα απλώς για να ακολουθηθούν οι διαδικασίες και είτε ε, υποβάλλουν έτοιμα ασύλου είτε επαναπροεθούνται. Αυτό μας είχε πει. Το ίδιο συμβαίνει στη Βουλγαρία. Θα ήθελα να γνωρίζω. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κύριος Μόραες, κύριε Ήλτσεφ, μπορείτε να απαντήσετε. Πάνω κάτω αυτό συμβαίνει και στη Βουλγαρία. Υπάρχουν κάποιες ιδέες, ίσως όχι εξαιρετικά καινοτόμε, αλλά σίγουρα χρήσιμες και οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, εγώ πρότεινα στις τουρκικές αρχές να υπάρχουν μικτές περιπολίες αξιωματικών της Frontex και του τουρκικού στρατού, οι οποίες θα φροντίζουν για την προστασία του συνόρου από την πλευρά της Τουρκίας. Δεύτερον, η παρακολούθηση προφανώς δεν είναι πρόληψη. Δεν μπορεί να σταματήσουμε έναν άνθρωπο να περάσει τα σύνορα απλώς και μόνο τοποθετώντας μια κάμερα. Αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στα σύνορα ακριβώ στη γραμμή τη συνοριακή, μπορούμε να τους δώσουμε πληροφορίες, μπορούμε να τους συμβουλέψουμε, κάτι που δεν γίνεται. Τώρα, επίσης φαίνεται ότι κάτι μας κρύβουν οι αρχές Τη ε, Τουρκία και της Ελλάδας. Τώρα δεν θα ήθελα να κατηγορήσω κανέναν, αλλά σοβαροί άνθρωποι, σοβαροί αναλυτέ μας λένε ότι υπάρχει το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων. Είναι εντυπωσιακό το γεγονό ότι οι άνθρωποι έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου, την άλλη άκρη της Μικράς Ασίας και φτάνουν στα ελληνοτουρκικά ή στα βουλγαροτουρκικά σύνορα και γνωρίζουν ακριβώς που είναι το πέρασμα. Δεν είναι εκπληκτικό αυτό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υποτιμήσουμε τις δυνατότητες και τις, ε, δυνατότητες που έχουν στα χέρια τους οι φίλοι μα από την Τουρκία. Εάν οι τουρκικέ αρχέ αποφασίσουν ότι έχουν τη βούληση να επηρεάσουν αυτέ τι μεταναστευτικέ ροέ, μπορούν να το κάνουν. Διαφορετικά, θα συνεχιστεί η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση τη αύξηση τη μεταναστευτική ροή προ τη Βουλγαρία και μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπου χωρί να έχει η Βουλγαρία τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται λοιπόν να ασκηθεί πίεση από εμάς προς την Άγκυρα, νομίζω αυτό είναι απαραίτητο. Απάντησα στο ερώτημά σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση αυτού του σημείου της ημερησίας διάταξης και 15 λεπτά πιο νωρίς από ό,τι είχε γραφεί στην ημερησία διάταξη μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5. Που αναφέρεται την εξασφάλιση κοινού ψηλού επίπεδου ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση. Η συγητής είναι από τους πράσινους, κ. Σλάιτερ. Έχουν κατατεθεί τροπολογίες μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, αλλά πολλές. Ωστόσο δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα πώς θα κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των τριών ε, συναρμόδιων επιτροπών, δηλαδή της ΙΤΡΕ, της ΙΜΚΟ και της ΛΥΜΠΕ. Θα το συζητήσουμε αύριο στη συνάντηση συντονιστών, το οποίο ίσως οδηγήσει στην αναβολή της ψηφοφορίας στη ΛΥΜΠΕ μέχρι να επιληθεί το ζήτημα αυτό. Κύριε Φλούιτερ, λοιπόν, έχετε το λόγο πριν δώσουμε τη ε, δυνατότητα στους σκιώδεις και στους υπόλοιπους ε, βουλευτές να παρέμβουν. Κύριε Σλούιτερ. Ευχαριστώ, αλλά δεν βλέπω να είναι παρόντες όσοι συνάδελφοι είχαν υποβάλει τροπολογίες. Εκείνους ήθελα να επιφυνθώ. Ελπίζω ότι οι βοηθοί τους θα μεταφέρουν αυτά που θα έχω να πω. Φαίνεται πως δεν συμφωνούμε ακριβώς σε σχέση με τον ορισμό της ε, κρίσιμης υποδομής, δηλαδή ποιες ε, εταιρείες θα καλύπτονται από την ε, οδηγία αυτή και ποιες υποδομές θα θεωρηθούν κρίσιμες υπό το έννοια αυτής της οδηγίας. Έχουμε συζητήσει το θέμα με τον εισηγητή της ε, ήτρε του κ. Σουάμπ και εκείνος μου είπε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το θέμα της, του ορισμού της κρίσιμης υποδομής. Πολλοί βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούν ότι ίσως η Επιτροπή να το παράκανε συμπεριλαμβάνοντας στις κρίσιμες υποδομές κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ε, δίκτυα αποθήκευσης δεδομένων. Ωστόσο, ίσως πιστεύω είναι χρήσιμο να καλύπτονται υποδομές ε, cloud computing, γιατί παρόλο που αυτό δεν ήταν και τόσο ενδεδειγμένο, υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν αποθηκεύσει τα δεδομένα των ασθενών τους σε τέτοιες υποδομές. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις το συζητήσαμε στο Στρασβούργο. Ένα άλλο θέμα, το οποίο τίθεται με πολλές τροπολογίες, είναι το ζήτημα των σημείων επαφής. Πώς θα μεταβιβάζονται αυτές οι πληροφορίες με τρόπο ασφαλή. Νομίζω εδώ πρέπει να βρεθεί μια ορθή ε, διαδικασία από τεχνικής απόψεως και νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι συχνά δεν πρόκειται για προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα. Δεν μπορούν εύκολα αυτά τα δεδομένα να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ανάλογα με το ποιο είναι ο φορέα που υποβάλλει αυτέ τι αναφορέ, θα πρέπει να είναι διαφορετικέ οι απαιτήσει. Για παράδειγμα, αν έχουμε μια τράπεζα που, της οποία στο πληροφοριακό σύστημα υπέστη επίθεση και αυτό εντοπιστεί, η τράπεζα θα πρέπει να γνωρίζει ακριβώς ποιοι ε, πελάτες της απειλήθηκαν από αυτή την παραβίαση. Όμω, όταν αυτή η τράπεζα θα ενημερώσει άλλε τράπεζε για να προσέχουν και εκείνε, δεν χρειάζεται να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τη. Χρειάζεται λοιπόν να περιορίσουμε τα δεδομένα τα οποία ε, μεταδίδονται ε, στα απολύτω απαραίτητα. Τώρα, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι επέβαλαν ε, τροπολογίε στα γερμανικά και δεν μπορούσα να τη διαβάσω, ζητώ συγγνώμη για τις τροπολογίες μου στα αγγλικά και γαλλικά που μπορώ, πρέπει να πω ότι περίμενα περισσότερες λύσεις, άσκηση κριτικής ή κάποιες ιδέες ε, για την προσπάθειά μου να υποβάλω πιο αυστηρούς προεπεριορισμούς στις εταιρείες λογισμικού. Από ό,τι φαίνεται το δέχτηκαν οι συνάδελφοι, ελπίζω να σημαίνει η μη κατάθεση τροπολογιών ότι δέχονται τις προτάσεις μου και ότι δεν πρόκειται να καταψηφίσουν την πρόταση συνολικά. Εν πάση περιπτώσει παραμένω ανοιχτός σε μια συζήτηση από αυτού του θέματος. Κάτι ακόμα. Είναι ε, ποιο θα πρέπει να φορέσει προ τον οποίο θα απευθύνονται αυτέ οι πληροφορίε, θα αποστέλλονται αυτέ οι πληροφορίε συγητή θεωρεί ότι θα έπρεπε αυτό να γίνεται μέσω των σημείων επαφή, αλλά υπάρχει και το πρόβλημα ότι ήδη έχουν υλοποιηθεί κάποια συστήματα, ήδη λειτουργούν αποτελεσματικά και ε, δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Τώρα είναι καλή ιδέα το να υπάρχει ένα μεμονωμένο, μοναδικό σημείο επαφή, υπάρχει καλύτερη διαφάνεια, αλλά δεν θα πρέπει να ε, καταστρέψουμε συστήματα τα οποία ήδη έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους ε, σήμερα. Άρα πρέπει να βρούμε μια συμβαστική λύση. Και εκεί υπάρχει μια τροπολογία από τον κύριο Άγκης για το ζήτημα. Είναι η τροπολογία 31 για το ζήτημα της αρμόδιας ε, πολιτικής αρχής σε εθνικό επίπεδο. νομίζω ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε το ρόλο αυτής της εθνικής αρχής. Αυτά από εμένα θα ήθελα να ακούσω και τους συναδέλφους. Ο πρόεδρος διαπιστώνω ότι δεν είναι όλοι εδώ παρόντες, αλλά η κυρία Χάνκης Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα Ουγγρικά για να ε, είμαι και πιο σύντομη. Και να σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα της διαπραγμάτευσής σας μέχρι σήμερα από την πλευρά του ΕΛΚ. Έχουμε υποβάλει τέσσερις τροπολογίες και θα μιλήσω μόνο εκπροσωπώντας τον εαυτό μου ε, και να πω ότι ευχαριστώ τον εισηγετή γιατί θα υποβάλει 30 τροπολογίες προσωπικά και στις 19 συμφωνήσαμε. Είναι ε, εξαιρετικό γεγονό ότι μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε τόσο πολλά θέματα τόσο νωρί. Εγώ θα εστιάσω στα θέματα εκείνα στα οποία υπήρξε συμφωνία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Το πρώτο είναι το ζήτημα του ορισμού της κρίσιμης υποδομής. Κρίσιμη υποδομή δηλαδή που μπορεί να αποτελήσει ε, αντικείμενο κυβερνοεπιθέσεων ή, ή ε, ηλεκτρονικής Εδώ προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική προστασία αυτής της κρίσιμη υποδομή. Δεν διαφωνεί κανένα αυτό, νομίζω. Αλλά συγκεκριμένα τι καλύπτει ο όρο κρίσιμε υποδομέ, νομίζω και εδώ συμφωνούμε στο ότι δεν θα πρέπει να είναι εξαιρετικά περιορισμό, περιοριστικός αυτός ο ορισμός, δηλαδή να μην αναφερόμαστε μόνο στις μεγάλες υποδομές. Θα πρέπει να υπάρχει υψηλή προστασία και σε άλλα συστήματα, όπως για παράδειγμα τα συστήματα διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου ή του δικτύου ίδρευσης ή της διαχείρισης της κυκλοφορίας γιατί αυτά τα συστήματα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Μια ηλεκτρονική επίθεση εναντίον αυτών των συστημάτων θα είχε τεράστιες επιπτώσεις για, στην καθημερινότητά μας και στην ασφάλειά μας, αν θέλετε. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να τονίσω το και θεωρώ σημαντικό είναι τα συστήματα cloud, τα συστήματα τα τα οποία μπορούν να υποστούν ε, επιθέσεις αρκετά πιο περίπλοκες, ε, phishing ή άλλου είδους. Ε, γι' αυτό από πλευράς προστασίας δεδομένων, πολιτικής προστασίας δεδομένων, εδώ το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για εξαιρετικά πολλά δεδομένα. είναι μαζική η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σε τέτοια συστήματα. Επομένω, θα πρέπει να βρούμε μια ε, προσέγγιση ισορροπημένη που θα εξασφαλίζει την προστασία αυτών των συστημάτων. Κάτι ακόμα και θα συνεχίσω. Ε, που έχει σχέση με την ε, ενίσχυση της ε, συνεργασίας. Θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των δημοσίων φορέων και των ιδιωτικών φορέων. Έχει υποβάλει ο συνάδελφο κ. Σόγκαν μια τροπολογία που έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα κατά την άποψή μου. Ζητάει από την Επιτροπή να καταγράψει και να συλλέξει όλες τις στρατηγικές ασφαλείας πληροφοριών των εθνικών αρμόδιων αρχών. Αυτό θα βοηθήσει τον συντονισμό και τη συνεργασία μας σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω έχουμε, συνολικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συμφωνήσει σε πολλά θέματα. Να επισημάνω και ένα στο οποίο ακόμα συνεχίζουμε τη συζήτηση και δεν ξέρω ακριβώ πού καταλήξαμε, αν συμφωνήσαμε ή όχι. Έχει υποβληθεί μια πρόταση που λέει ότι ίσως θα πρέπει να περιμένουμε την, τον νέο κανονισμό για την προστασία δεδομένων και να μην ψηφίσουμε αυτή την, αυτή την ε, απόφαση πριν ε, εγκριθεί αυτός ο κανονισμός. Το ΕΛΚ ε, δεν θα συμφωνούσε με μια τέτοια προσέγγιση. Ο κύριος Φάμπ έχει υποβάλει διάφορα στροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στην προστασία προσωπικών δεδομένων και αυτές οι τροπολογίε θα μας δώσουν την ευκαιρία να ενισχύσουμε το επίπεδο προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το θέμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και σημαντικό, επομένως οποτεδήποτε έχουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε την προστασία ε, των προσωπικών δεδομένων, οποτεδήποτε έχουμε αυτή τη δυνατότητα, το ΕΛΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Γιατί λοιπόν να αναβάλουμε την έκθεσή μας, αντιθέτως πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Η κυρία Φάιρ δεν είναι παρούσα. Για τους σοσιαλιστές δεν βλέπω κάποιον να θέλει να πάρει το λόγο. Εξ ονόματος τώρα των φιλελευθέρων. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Χάνκης. Πιστεύω ότι είναι λίγο παράδοξο το ότι από τη μια το Συμβούλιο ζητάει αναβολή του πακέτου μέχρι το 15 ή και πέραν το 2015. Αν κάτι τέτοιο επιθυμεί το Συμβούλιο, αν θέλει να περάσει αυτή η, το πακέτο προστασίας, δεν μπορεί να αναβάλει αυτή την ψηφοφορία. Το Συμβούλιο πρέπει να συγκροτηθεί και να καταλάβει ότι αυτό έχει άμεση σχέση και με την προστασία ε, των δεδομένων. Μου φαίνεται λοιπόν παράδοξο το γεγονός ότι από τη μία αναφερόμαστε σε κάποιες επιθέσεις ε, από μέρους κάποιων ε, τρομοκρατών, κακών και από την άλλη αυτός ο οποίος έχει πρόσβαση στα συστήματά μας είναι ο καλύτερος μας φίλος αυτοί που προετοίμαζαν αυτά τα κείμενα δεν φανταζόταν ότι αυτός ο οποίος θα κατασκοπεύσει είναι οι Αμερικανοί, οι φιλικές χώρες, συμμαχικές χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να πω εδώ ότι εάν μια τέτοια επίθεση λάβει χώρα από μια ξένη χώρα, παραδείγματος χάρη στην Ολλανδία, στη Ολλανδία η οποία όντως υπέστη τέτοιες ε, επιθέσεις στο σύστημα και ξέρουμε τι έγινε με το SWIFT. Το ίδιο έγινε και στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο έγιναν μαζικές παραβιάσεις. Η αντίδραση ποια ήταν, ξέρω τι συνέβη στην Ολλανδία, δεν ξέρω για το Βέλγιο, τίποτα. Και θα πρέπει ίσως να ξαναδούμε το πώς μπορούμε να αμυνθούμε τι καταρχήν διερεύνηση αποφασίζεται να γίνει. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο να είμαστε 27 κράτη που δεν μπορούμε να αποφασίσουμε να διερευνήσουμε και οι μόνοι που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο είναι η Europol. Ποιοι είναι οι άλλοι οι και όδης για το ECR. Δεν είναι ακόμα δηλαδή και αν το θέμα αυτό ε, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί ερχόταν στην ημερήσια διάταξη στις 5. Η κυρία Βερζά επίσης δεν είναι παρούσα. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Συμφωνώ μαζί σου. γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μάθαμε κάποια πράγματα που ήταν γνωστά από τον Ιούνιο βεβαίως ότι περίπου τα δεδομένα τριών εκατομμυρίων ασθενών από τη Σουηδία βρισκόταν κάπου και βεβαίως υπήρχε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, κάτι το οποίο είναι μια σαφής παραβίαση αυτού που ορίζει αυτή η οδηγία. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και από μέρους των υπηρεσιών ασφαλείας ε, όσον αφορά τις παραβιάσεις ε, της ε, προστασίας των δεδομένων. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε τόσο αφελείς. Εγώ θυμάμαι πριν από τρία χρόνια τις διαπιστώσεις που είχαν γίνει και το πόσο μας καθησύχασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αν σήμερα γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευθούν σε ένα cloud και η πρόσβαση είναι τόσο εύκολη Καταλαβαίνετε ότι αυτό που μπορεί να μας προστατεύσει δεν είναι κανονισμοί και ρυθμίσεις όταν ξέρουμε ότι από τεχνικής απόψεως είναι ευάλωτα τα συστήματα. Το ίδιο μπορεί να πει κανεί και με τις τηλεφωνικές ε, συνδιαλέξεις. Απορώ παραδείγματος χάρη πως η Γερμανίδα Καγκελάριος ε, δεν είχε ένα σύστημα το οποίο να την προστατεύει στο τηλέφωνό της. Αυτό που είπε η Άνια Είναι σωστό ότι τις περισσότερες φορές οι παραβιάσεις δεν είναι ε, σκόπιμες. Πρόκειται για τεχνικά ή ανθρώπινα σφάλματα ή λανθασμένες ή κακές διαδικασίες. Τώρα, για όλες τις ε, υπόλοιπες παραβιάσεις ε, δεν ξέρω αν υπάρχει σύστημα αποτελεσματικό για να μας προστατεύσει και να προστατεύσει και τα δεδομένα μας. Για την Europal δεν ξέρω ποια είναι η θέση ούτε της ε, ομάδας μου, αλλά ούτε εγώ το έχω σκεφτεί. Θα περιμένουμε να δει τι θα πει η Άνια. Πρόεδρος, το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δική μου έκθεση που είναι η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Και αυτό αφορά βεβαίως το σύστημα PNR, τα δεδομένα των επιβατών. Κοιτώ το ρολόι, κοιτώ και πώς είναι παρόντες στην αίθουσα. Α, κάποιος μπήκε. Και για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Δεν έχω προετοιμάσει ακόμα κανένα σχέδιο έκθεσης. Είχαμε παρακολουθήσει μία κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση πριν από 7 μήνες μας παρουσίασε η Επιτροπή τότε την κατάσταση, είχαμε υποβάλει κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί ακόμα, ικανοποιητικά τουλάχιστον. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ μίλαμε για μια συμφωνία με τον Καναδά και δεν έχουμε καμία απολύτως ε, εγγύηση ότι τα δεδομένα τα οποία μπορούμε εμείς να παρέχουμε στον Καναδά δεν θα διαχειθούν μέσω συμφωνιών που έχει ο Καναδάς με άλλες χώρες παντού στον πλανήτη. Προτίθεμε λοιπόν να αναβάλουμε αυτή τη στιγμή τη συζήτηση μέχρι να υπάρξει μια ε, έκκληση για συμφωνία. Ο κύριος Λίτερ όμως ζητάει το λόγο. Κοιτάξτε, βεβαίως μπορείτε εσείς να επιλέξετε πώς θα προχωρήσετε. Το θέμα είναι όμως ότι από τη στιγμή που έχουμε συμφωνίες στο παρελθόν, οι οποίες σήμερα είναι αντικείμενο τέτοιες κριτικής, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να προσέχουμε. Ναι, Πρόεδρος, με την ίδια ε, λογική, με αυτό που κάναμε το 2010 στην προηγούμενη συμφωνία, υπήρχε ένας κατάλογος κριτηρίων και αυτό βεβαίως υπάρχει και ισχύει για πολλές συμφωνίες και είναι ένας κατάλογος κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε υποβάλει ερωτήσεις από το 2009 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και απαντήσεις δεν έχουμε λάβει. Αν θέλει λοιπόν η συμφωνία η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει απαντώντας αυτές τις ερωτήσεις. Και βεβαίως τι γίνεται με τις συμφωνίες μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών στην προκειμένη περίπτωση. Συμφωνείτε όλοι να μην συζητηθεί το θέμα τώρα, ωραία. Και αν δεν υπάρχουν και άλλες παρατηρήσεις, ολοκληρώθηκε η συνεδρίασή μας για σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ.